Καλησπέρα σας. Με ακούτε παρακαλώ. Όχι, μάλλον. Λοιπόν, καλώς ορίσατε όλοι στην απογευματινή μας ε, συνεδρίαση. Αντικαθιστώ τον πρόεδρο της Επιτροπής Προπολογισμών, αλλά αυτό είναι καλό μόνο για τη διερμηνία. So, uh, this is not working in Χρησιμοποιήστε παρακαλώ τα ακουστικά. Είναι η μόνη λύση και πάλι καλώς ορίσατε στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών ε, με την Επιτροπή ΕΚΟΝ για να μιλήσουμε για το πρόγραμμα στήριξης μεταρρυθμίσεων. Έχουμε και ανακοινώσει ε, για τον προϋπολογισμό. Υποθέτω ότι είναι αποδεκτή η μερσή διάταξη, δεν είναι επίμαχη. Έχουμε μόνο 45 λεπτά στη διάθεσή μας και στη συνέχεια θα συνεδριάσουν ξεχωριστά οι δύο επιτροπές. Περνώ λοιπόν κατευθείαν στο σημείο 3 που είναι το πρόγραμμα στήριξης μεταρρυθμίσεων. Και καθώς έχουμε μόνο 45 λεπτά, πρέπει να θέσω και χρόνο ομιλίας για τους ομιλητές. 5 λεπτά για τους εισηγητές, τους έχουμε εδώ στην αίθουσα και τους δύο. Και θα ξεκινήσουμε με την Άιντερ Γουάρντα Σαμπάλ για να συνεχίσουμε τα όσα συζητήσαμε από την προηγούμενη συνεδρία. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω μάλιστα να ξεκονομήσω και χρόνο. Καταρχήν, θέλω να εξηγήσω γιατί κάνουμε αυτή τη μεικτή συνεδρίαση αυτή τη στιγμή καθώς ε, δεν έχουμε ως εισηγητές να παρουσιάσουμε κάτι στις επιτροπές αυτή τη στιγμή, αλλά μας φάνηκε καλό να ενημερώσουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, όχι για τις διαπραγματεύσεις, ε, αλλά για τις συζητήσεις ε, που υλοποιούμε για το πρόγραμμα στήριξης μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων και να εξηγήσουμε τις αλλαγές που παρουσιάζει το Συμβούλιο έτσι ώστε να έχουν όλοι την ίδια εικόνα. Parece que tenemos algún problema con el sonido hoy. ό,τι έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον ήχο. Προετοιμάσαμε μια μικρή σύνοψη για να τα έχετε και γραπτός και να παρακολουθείτε τις εξηγήσεις μας. Και τα βλέπετε στην οθόνη. Το πρώτο τμήμα θα δείτε όλα τα βήματα που έχουν γίνει και γιατί αυτή τη στιγμή συζητούμε την πρόταση αυτή. Τώρα φαίνεται ότι λειτουργεί. Bueno, Όπως ξέρετε, Δύο χρόνια έχουμε επιτάπητο στην πρόταση αυτή. Πρόκειται για μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτή η Επιτροπή και η Επιτροπή Προπολογισμών αρχίσαμε να εργαζόμαστε επί της ανάγνωσης, αλλά παράλληλα με τις εργασίες στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο άρχισε τη δική του εξέταση. Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, αυτό που γνωρίζαμε ως πρόγραμμα στήριξης μεταρρυθμίσεων εξελίχθηκε προς πρόγραμμα στήριξης μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων και μάλιστα προσθέθηκε αυτό το νέο μέσο το δημοσιονομικό για την ανταγωνιστικότητα και τη σύγκληση. Δυστυχώ δεν μπορέσαμε να φτάσουμε σε κοινή θέση στην προηγούμενη θητεία στο Κοινοβούλιο, όμως ε, είναι αλήθεια ότι και αν είχαμε φτάσει σε κοινή θέση δεν ε, θα μπορούσε να υλοποιηθεί γιατί θα είχαμε βασιστεί στο κείμενο που παρουσίασε η Κομισιόν και που αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει οριστικά από τις διάφορες προεδρίες. Έχει αλλάξει εντελώ. Αυτή τη στιγμή επισήμως έχουμε μόνο μία πρόταση επιτάπητος της Φιλανδικής Προεδρίας. Όμως γνωρίζουμε ότι και η Κροατική Προεδρία όπως και η αρμόδια ομάδα εργασίας στο Συμβούλιο εργάζονται επί κάποιων πτυχών και ακόμη δεν έχει υπάρξει συμφωνία. Ως εισηγητές εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από την θέση της Κροατικής Προεδρίας για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και την εργασία στις επιτροπές μας. Όχι γιατί θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτό που θα έρθει από το Συμβουλίο, αλλά γιατί δεν θα είχε νόημα να εργαστούμε επί ενός εγγράφου που δεν ε, έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο. Δεν θέλουμε δηλαδή να εργαζόμαστε μάταια. Επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, για να σας εξηγήσω τις διάφορες αλλαγές από την πρόταση που είχαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως την τελευταία πρόταση που έχουμε επιτάπητος. Ξέρετε ότι στην πρόταση της Κομισιόν είχαμε τρία μέσα, το Reform Delivery Tool, το Convergence Facility και το Technical Support. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ε, Πάλι έχουμε τρία μέσα, η τεχνική υποστήριξη συνεχίζει να είναι η ίδια, όμως το εργαλείο ε, για την παράδοση των μεταρρυθμίσεων όπως συμμετείχαν μέλη της Ευρωζώνης ε, και μέλη εκτός Ευρωζώνης τώρα διαιρείται σε δύο μέρη. Συγγνώμη γιατί είναι κάπως πολύπλοκο να το εξηγήσω, αν ε, και με το γράφημα νομίζω θα τα καταλάβετε καλύτερα. Επομένως έχουμε ένα πρώτο εργαλείο που είναι το εργαλείο ανταγωνιστικότητας και σύγκλησης που τώρα βασικά θα απευθύνεται στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και το τμήμα που αφορά τα κράτη-μέλη που δεν είναι στο Ευρωζώνη και που αφορά τη σύγκληση μετατρέπεται σε ένα νέο εργαλείο που αφορά τα κράτη-μέλη που είναι εκτός Ευρωζώνης και που θα ονομάζεται τώρα Μέσο για τις μεταρρυθμίσεις και τη σύγκληση. Και όπως είπα πριν, το μέσο τεχνικής υποστήριξης συνεχίζει το ίδιο. Αυτή είναι η πρόταση που έχουμε επιτάπητο αυτή τη στιγμή και από την πλευρά της Φιλανδικής Προεδρίας, δηλαδή επίσημη πρόταση, όπως και της κρατικής Προεδρίας. Όμως ακόμη δεν έχουμε ενημέρωση για τις τροποποιήσεις. Και θα δώσω το λόγο στο συνεισηγητή. Όμως, να σας πω ότι στην τελευταία πρόταση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τα δις δηλαδή, που αρχικά είχε παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Φυσικά αυτό θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο την επόμενη Πέμπτη στο Συμβούλιο, αλλά όλα τα νούμερα που έχουμε επιτάπητος είναι κάτω από τα 25 δισεκατομμύρια που αρχικά είχαν προταθεί. Νομίζω ότι ξεπέρασε τα 5 λεπτά, αλλά ήταν κάπως πολύπλοκες οι εξηγήσει και θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο. Oh, Ευχαριστώ, Άιντερ. Δεν υπάρχει συνέχεια στους συζητητές από την ΕΚΟΝ και γι' αυτό έχουμε το Ρενιού, τον κύριο Πισλάρο. Εισηγητή για το ίδιο ζήτημα. Έχετε πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Με χαρά σας αναφέρω ότι καταρχάς έχουμε μια πολύ καλή ομάδα με την Άιντερ, Κάρντια, Θαμπάλ και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς στις διαδικασίες μας, θέλουμε να πετύχουμε να καταλήξουμε σε μία θέση για το Κοινοβούλιο. Από τη στιγμή που ο φάκελος αυτός έχει αλλάξει τόσο πολύ, κάτι που το είπε και η συνάδελφος. Στην παρουσίαση του PowerPoint έχουμε κάποια πράγματα που σας δίνουν τη δομή της συζήτησης. Είναι δύσκολο να το παρακολουθήσει κανείς γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι και η τελευταία μορφή εμπασχευτός του κειμένου, αλλά βασιζόμαστε στη φιλανδική πρόταση. Και τα κεφάλαια που εξετάζουμε έχουν να κάνουν με τη νομική βάση και την επιλεξιμότητα. Και βλέπετε και τα τρία βασικά που βλέπουμε. Άρα έχουμε μια νομική βάση με συμμοχή για το δημοσιονομικό εργαλείο για τη σύγκληση και την αντιαγωνιστικότητα και ασχολούμαστε επίσης με τις μεταρρυθμίσεις, τις χρηματοπιστωτικές και για το ΚΡΙ, το ε, Εργαλείο Σύγκλησης και Μεταρρύθμισης. Βλέπετε περί πρόκειται και για τις ε, χώρες που είναι σε διαδικασία ένταξης και έχουμε και την τεχνική στήριξη που βασίζεται στο εργαλείο του ε, συστήματος για τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων SRSS, SRSP. Τώρα η διακυβέρνηση και οι διαδικασίες ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Βασιζόμαστε στο, στο Eurogroup και στο Euro Group Έχουμε τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης, ε, βασιζόμαστε στα CSR και στα NRP. Ε, διαφοροποιούμε ανάλογα με το εργαλείο. Ένα άλλο θέμα που μας ενδιαφέρει είναι η κατανομή των ε, κονδυλίων. Βλέπουμε ότι εισάγεται εδώ ένα νέο κριτήριο με το ΑΕΠ, το κατακεφαλήν εισόδημα, το αντίστροφο δηλαδή αυτού. Και καλούμε όλους να μπουν σε αυτή τη συζήτηση μαζί μας. Υπάρχει και το θέμα του προϋπολογισμού με τα 25 δις για τα οποία γίνεται λόγος. Έχει ήδη τονιστεί. Να σταθώ λίγο στο γεγονός ότι υπάρχει αυτό το εργαλείο. Μπορούν τα κρατημέλη και για την τεχνική στήριξη να φτάσουν σε top-up, σε κατόφλια με τις διακυβερνητικές συμφωνίες και μετά να έχουμε θελούσια μεταφορά για περαιτέρω ζητήματα τεχνικής στήριξης. Άρα ο προπολογισμό αποτελείται από τον προπολογισμό του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου συν αυτού που θα εισφέρουν τα κράτη-μέλη αυτά καθε αυτά. Δύο λόγια για το χρονοδιάγραμμα. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εξαρτόμαστε από τις συσκέψεις και συνεδριάσεις στις 17 και στις 20 του μηνός. Έχουμε τη συνεδρίαση του Eurogroup. Άρα η αρχική μας καταληκτική προθεσμία ήταν να αποσταλεί το σχέδιο έκθεσης στις 2 Μαρτίου, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατό. Είχαμε την πράσινη εβδομάδα Και δεν ήταν πολύ δημοφιλές αυτό, γιατί ρώτησα εδώ και δεν υπήρχε μεγάλη βούληση. Άρα, με τη βοήθεια της γραμματείας, την οποία θέλω να ευχαριστήσω θερμά, παρατείνουμε την καταληκτική προθεσμία, καταληκτική ημερομηνία για την 20η Μαρτίου και θέλουμε στις 21 Απριλίου να είναι η καταληκτική προθεσμία ημερομηνία για την παρουσίαση της έκθεσης. Ε, υπάρχουν κάποιες φήμες που κυκλοφορούν στους διαδρόμους και θέλω να τις διασαφίσω. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών είναι πολύ μικρή, είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα ε, εν ώψη της 21ης Απριλίου και θα το αλλάξουμε αυτό για να έχει κάθε επιτροπή του Κοινοβουλίου μία εβδομάδα ε, διάθεση και περιθώριο για τροπολογίες. Μετά θα εξεταστούν οι τροπολογίες 27 και 28 Μαΐου και θα ψηφιστεί ε, στην Επιτροπή 27 και 28 Μαΐου και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Ιουνίου είτε την πρώτη είτε τη δεύτερη. Ελπίζουμε ότι αυτή η πολύ σημαντική μεταρρύθμιση θα ληφθεί πολύ προσεκτικά υπόψη με σοβαρότητα από το Συμβούλιο, με τη σοβαρότητα που της αξίζει και που της αναλογεί. Ελπίζουμε να φτάσουμε γρήγορα σε μια κοινή θέση, έτσι ώστε αυτό το έγγραφο, το τόσο σημαντικό για τα κράτη-μέλη και για τον Ευρωπαίο πολίτη, να μπορέσει να εκρηχθεί. Και θέλω να ολοκληρώσω κάπου εδώ ευχαριστώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεισφορά της και καλώντα της να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις, εάν το επιτρέψει βεβαίως ο Προεδρεύων στη δική μας συνεδρίαση της ε, Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής. Ευχαριστώ. Είμαι συμπρόεδρο με τον κύριο ε, Κοσμάο, γιατί είναι κοινή η συνεδρίαση, δεν το έχετε παρατηρήσει, με την Επιτροπή ΕΚΟΝ και την Επιτροπή Budget. Ο κύριος Κύρτσος νομίζω έχει ζητήσει το λόγο, αλλά νομίζω ότι δεν είναι στην αίθουσα και γι' αυτό στρέφομαι στην κυρία ε, Μάικλ. Σκιώδης για το ΕΛΚ. Δύο λεπτά, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ και θα είμαι το συντομότερο. Θα είμαι όσο δυνατόν συντομότερο. Εκπροσωπώ τον κύριο Καράς, ε, που ήταν ο εισηγητής του ΕΛΚ για το RSP, για το πρόγραμμα στήριξη μεταρρυθμίσεων. Έχει κάποιες κατεπίγουσες υποχρεώσεις, γι' αυτό δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Πέντε σημεία έχω να αναφέρω. Πέντε. Καταρχάς, ο κύριος Κάρας υποστηρίζει τον συνολικό απότερο στόχο αμα, του προγράμματος στήριξη μεταρρυθμίσεων, όπως αναφέρθηκε να υποστηριχθεί η υλοποίηση των διευθυντικών μεταρρυθμίσεων προτεραιότητα σε όλα τα κράτη-μέλη και εκ παραλλήλου να ενισχυθούν οι επενδύσεις και να υπάρχει σωστή και υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. Οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν τμήμα αυτού του ενάρτου τριγώνου στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμένου. Και αυτό θα πρέπει να γίνει όταν τα κράτη-μέλη έχουν υλοποιήσει κατά μέσο όρο 53% της ε, ε, συστάσεις μεταξύ του 2012 και τώρα. Και αυτό σημαίνει 1% μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κατανοήσουμε και την κλίμακα του εργαλείου αυτού για τις επενδύσεις στο μέλλον και την ενδεχόμενη υψηλή απόδοση. Εκ παραλλήλου, αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί τμήμα της εμβάθυνσης που είναι απαραίτητη σε ό,τι αφορά την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν να καταβάλουμε προσπάθειες. Κατά δεύτερον, ο κύριος Κάρας καλώς ορίζει το γεγονός ότι η διαπραγματευτική ομάδα στην διαδικασία αυτή θα εξετάσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πλαίσιο διακυβέρνησης για το δημοσιονομικό μέση, για τη σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα που βασίζεται στις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο, αλλά το Κοινοβούλιο είναι συνομοθετή. Επίσης, όρος. Και δεν πρόκειται λοιπόν να κάνουμε copy-paste των όρων που θα συμφωνηθούν. Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε του καλύτερου δυνατού στόχου προ το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Πέρα και από αυτά που είχε κάνει το Κοινοβούλιο στην προηγούμενη θητεία. Τρίτον και πολύ σύντομα, ο κύριο Κάρας υποστηρίζει τη δημιουργία ειδική δυνατότητα για την υποστήριξη για τεχνική και δημοσιονομική σύγκληση για χώρε που δεν είναι στο ευρώ προ τον χώρο του ευρώ, όπω είχε ήδη προτείνει και η Επιτροπή Juncker. Τέταρτον, ο κύριος Κάρος υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε άνηση υποστήριξη των ε, μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να αποφευθεί και θα πρέπει ο μηχανισμός εξάντα επίση να λειτουργήσει σωστά και να σχεδιαστεί σωστά. Τελευταίο στοιχείο, ο κύριο Κάρα θέλει να υπογραμμίσει ότι το εργαλείο αυτό θα πρέπει να συνάδει και με την μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης, επί της οποίας έχει υποβάλει προσφατώς ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, ο κύριος Κάρας δεν θα υποστηρίξει την διενέργεια ε, τέτοιες αναθεωρήσεις για το θέμα αυτό, γιατί αυτές οι δύο πρωτοβουλίες θα πρέπει να προχωρήσουν και να συμπληρώσουν η μία την άλλη, όχι να αντικαταστήσουν και να εμποδίσουν η μία την άλλη. Προκειμένου λοιπόν να επιληθούν όλα αυτά τα ζητήματα, ο κ. Κάρας προσβλέπει στη συνεργασία με τους συνεισηγητές και με όλη την ομάδα διαπραγμάτευσης της Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή δεν έχουμε, μάλλον επειδή δεν έχουμε άλλον συντονιστή από το ΕΛΚ, σα έδωσα παραπάνω χρόνο και σε ό,τι αφορά και την προσάρτηση στην Ευρωζώνη. Να περάσουμε τώρα στου σοσιαλιστέ και δημοκράτε. Αλλά διαπιστώνω και πάλι απουσία του σκιώδη του σοσιαλιστών και δημοκρατών ε, από το Ρινιού τώρα, κύριο Γκαρικάνο, αν ε, και εφόσον είναι εδώ. Μα φαίνεται η Δευτέρα είναι δύσκολη ημέρα για αυτές τις κοινέ συνεδριάσεις. Και το idea που σιάζει. Και έτσι κερδίσουμε πολύ χρόνο σε ό,τι αφορά το χρόνο ομιλία των σκιωδών. Από τους πράσινους τώρα, κύριος Μπεσλάγκερ. Ναι, εδώ είμαι. Ναι, και εγώ εκπροσωπώ τον, ε, επίσης και τον σκιώδη της Επιτροπής Εικόν για να τα παρουσιάσω όλα αυτά πιο συνοπτικά. Καταρχάς, χαίρομαι που έχουμε αυτή την αναλλαγή απόψεων. Και επειδή δεν υπάρχει ακόμα νομική βάση να εξετάσουμε, θα επικεντρωθώ στην πρόσφατη πρόταση που είδαμε από την Προεδρία στο διαπραγματευτικό αυτό κουτί. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, ευελιξία, έχω τρία στοιχεία να αναφέρω. Κοιτώντα τα θέματα διακυβέρνηση. Το διαπραγματευτικό κουτί φαίνεται να έχει αυτή την ε, φιλοδοξία ότι θα πρέπει να μπουν αυτά τα ζητήματα στο στρατηγικό προπολογισμό των κρατών μελών. Ξέρουμε ότι το πρόγραμμα στο ΔΕΛΤΑΠΗ δεν είναι επιπρόσθετο, αλλά ουσιαστικά αφαιρεί χρήματα από υφιστάμενα προγράμματα και έργα. Και άρα ουσιαστικά αυτά τα χρήματα, αυτά τα κονδύλια θα αφαιρεθούν από το τομεί όπου ισχύει συναπόφαση για το Κοινοβούλιο και θα δαπανηθούν σε άλλου τομεί και άλλε μορφέ διακυβέρνηση όπου θεωρούμε ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνεια και δεν υπάρχει σε κάθε περίπτωση συναπόφαση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί να συμφωνήσει το Κοινοβούλιο σε αυτή την εναλλακτική διάσταση των πόρων σε διακυβερνητικό επίπεδο. Κατά δεύτερον, και πάλι έχει μειωθεί ο όγκος. 25 δις ε, ήταν η αρχική πρόταση, η τελευταία πρόταση όμως τώρα προτείνει να υπάρξει ένα δημοσιονομικό εργαλείο με πολύ περιορισμένη δημοσιονομική ικανότητα αλλά τεράστια θέματα διακυβέρνηση. Γιατί να υποστηρίξουμε λοιπόν το εργαλείο αυτό. Δεν καταλαβαίνω το οικονομικό όφελο, το πολιτικό όφελο ενό τέτοιου εργαλείου. Εκτό και αν έχουμε επιλύσει τα θέματα και σε ό,τι αφορά το ύψο ε, του εργαλείου και τη διακυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τώρα την ευελιξία, έχω ένα τρίτο σχόλιο. η λογική η οποία μας προβλημάτιζε δεν βλέπουμε να έχει, μάλλον έχει αφαιρεθεί, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον θα ανακύψει εκ νέου σε, σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που μας ανησυχούν, σε ό,τι αφορά δηλαδή τη διαμόρφωση αυτού του δημοσιονομικού εργαλείου κατά τρόπο που να μας ικανοποιεί. Τέταρτο σχόλιο και τελευταίο, το CRI και τα στρατηγικά κεφάλαια και κονδύλια δεν είμαι σίγουρη πως θα διευθυνθούν. Ως τώρα ισχύει το σύστημα κατακεφαλής ε, ΑΕΠ και δεν βλέπω γιατί να μην ισχύει το ίδιο και στο Ταμείο Συνοχής. Και κατά δεύτερον πιστεύω ότι το... η κλίμακα του εργαλείου είναι αρκετά μεγάλη σε ό,τι αφορά το συνολικό πακέτο. Θα θέλαμε λοιπόν να μας εξηγήσετε γιατί υπάρχει τέτοια διαμόρφωση σε ό,τι αφορά τις χώρες στόχο. Αυτά ήταν τα σχολεία που είχα σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο πιο πολύ, όχι τόσο το χρονοδιάγραμμα. Ελπίζω να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά και σαφώ να αποστείλουμε ω μήνυμα προ το Συμβούλιο ότι δεν πρέπει να αποτεχτούμε τυφλά τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Για να δούμε τώρα. Θέλουμε να δούμε αν είναι εδώ οι ε, του ECR. Ο ένας λείπει, ο άλλος όμως ε, μπορεί να χαλαρώσει λίγο. Για να δούμε ο κύριος Ροπετζήλη είναι εδώ. Μάλιστα. Για να δούμε αν είναι εδώ τώρα η Σκιώδης από την ΚΟΥ, ο κύριος Παπαδημούλης. Όχι. Αλλά ευτυχώ ο γείτονα μου είναι εδώ, ο κύριος Γκουσμάου. Σκιώδης για την ΕΚΟΝ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω πρωτογαλλικά. Το θέμα που έχει να κάνει με το πρόγραμμα στήριξης διορθωτικών μεταρρυθμίσεων είναι να γνωρίζουμε ακριβώς αυτό γιατί δημιουργούμε αυτό το εργαλείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν ε, ο σκοπός είναι να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο αυτό για να παρακάψουμε το γεγονό οτι ότι πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν σεβαστεί τι συστάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπή να δημιουργήσουμε δηλαδή μια δημοσιονομική κατότητα που θα έχει ω στόχο να οθήσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τι διαφορετικέ ε, μεταρρυθμίσει που κάποιε κυβερνήσει θεώρησαν ότι είναι αντιπαραγωγικέ. Έτσι λοιπόν η συζήτηση για τι διαφορετικέ μεταρρυθμίσεις και η δυνατότητα να έχουμε δημοσιονομική ικανότητα για την Ευρωζώνη μα βάζει σε διαφορετικό επίπεδο με διαφορετικέ μεταρρυθμίσεις. Ουσιαστικά θα πρέπει να νομιμοποιούνται από τους ευρωπαϊκούς δημοκρατικούς θεσμούς και ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, τις Εθνικές Κυβερνήσεις κτλ. Και κατόπιν χρειαζόμαστε μια δημοσιονομική ικανότητα που ε, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός της Ευρωζώνης. Κάτι που φαίνεται δεν πρόκειται να κάνει το BIC, ε, ούτε σε ό,τι αφορά τον κανόνα ανακατανομή ούτε σε ό,τι αφορά τον όγκο του εργαλείου που χρειαζόμαστε. Ε, γιατί θα χρειαζόμασταν κάτι τεράστιο αν το συγκρίνουμε τις ανισορροπίες που έχουμε στην Ευρωζώνη. Έτσι λοιπόν, φυσικά εμείς θα συμμετάσχουμε στη συζήτηση αυτή και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα στήριξη μεταρρυθμίσεων και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τελικά σε τι θα χρησιμεύσει αυτό το μέσο και ποιο είναι ο βαθμός του ελέγχου και της δημοκρατικής νομοποίηση που θα έχουν οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Γιατί φυσικά αν αυτά αποφασιστούν μόνο από το Eurogroup και την Κομισιόν, εμεί δεν θα είμαστε υπέρ. Μάλιστα η χώρα του κυρίου Γκουσμάου έκανε τεράστια προσπάθεια να ξεπεράσει την κρίση χωρίς δημοσιονομικά κίνητρα ιδιαίτερα μεγάλα. Τώρα, έχουμε κάποια λεπτά για το κατσδιάι. Αν θέλει κάποιος να ζητήσει το λόγο, παρακαλώ. Τι έκπληξη. Ε, Αν ναι, όχι, κομισιόν. Α, συγγνώμη κύριε Σόντσα. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πολωνικά. Ο κύριος ε, Ρόμπερτ Σίλε αποσιάζει, αλλά εγώ είμαι ο δεύτερος ε, σκιώδης εισηγητής και καθώς ε, μας το επιτρέπει ο χρόνος θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η δική μου ομάδα είναι υπέρ της τεχνικής υποστήριξης. Αυτή είναι μια ιδέα που θα πρέπει να διατηρηθεί. Φυσικά όλα τα νέα μέσα τα οποία θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα, δεν τα καταδικάζουμε, δεν λέμε ότι πρόκειται για κάτι κακό, όμως είναι πολύπλοκη η κατάσταση. Υπάρχουν ε, κάποια κράτη που ανήκουν στην Ευρωζώνη, κάποια άλλα που δεν ανήκουν. Επομένως, η δική μας ομάδα θα παρουσιάσει μια πιο λεπτομερή θέση σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Όλα όσα αφορούν τον προπολογισμό μας ενδιαφέρουν. Ε, έχουμε τώρα μια νέα διαχείριση του προπολογισμού, τους ιδίους πόρους, όλα αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα για μας. Η πολωνική κυβέρνηση δεν διστάζει να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων αυτών και μάλιστα είναι έτοιμη να συνεισφέρει ακόμη περισσότερο σε αυτό το νέο προπολογισμό, γιατί μας ενδιαφέρει η συνοχή στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πιο φτωχές ε, μετακομμουνιστικές κόρες ε, θα πρέπει να συνεχίζουν να είναι σημαντικοί δικαιούχοι των ε, χρηματοοικονομικών μέσων που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η υποστήριξη είναι ιδιαίτερα ορατή σε αυτά τα κράτη. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι θα είναι και ισχυρή η φωνή μας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, συνεχίζεται και θα δούμε καταρχήν ποια θα είναι η θέση του Συμβουλίου και ποιος θα είναι και ο δημοσιονομικός φάκελος, ποιο θα είναι το ποσό. Βέβαια, θα λάβουμε υπόψη τι μας ε, ενδιαφέρει και τι μας συμφέρει ως Ένωση. κυρία Ζερλαντίν Μαγιού από την ΓΑΜΑ Μεταρρυθμίσεων, παρακαλώ. Είναι εδώ, ευτυχώς. Um, yes, ναι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που δίνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψή της. Εν μου ζητήσατε να σας πω πού βρισκόμαστε σε σχέση με τις τρέχουσες εξελίξεις. Συνεργαστήκαμε εντατικά με τη Φιλανδική Προεδρία, τώρα συνεργαζόμαστε με την Κροατική Προεδρία για να ενσωματώσουμε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που έχουν προβληθεί στο term sheet και να, τα, να τους βρούμε την κατάλληλη θέση. Να βρούμε την κατάλληλη θέση για τις αλλαγές αυτές στο, στο εφιστάμενο πρόγραμμα στήριξης. Το κείμενο της Φιλανδικής Προεδρίας το έχουμε μοιράσει, το έχουμε μοιραστεί μάλλον με τους δύο συνειζηγητές και αυτό αποτελεί μια σχετικά σταθερή βάση. Εξελίξεται η συζήτηση για το allocation process και για την αξιοποίηση των κονδυλίων με πιο ευέλικτο τρόπο, μέχρι το 20% βεβαίως. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι ακόμα υποσυζήτηση και ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση και να βοηθήσουμε την Κροατική Προεδρία να προχωρήσει τη φιλοδοξία της, το στόχο της που είναι να έχει ολοκληρωθεί η εξέταση μέχρι τα τέλη Μαρτίου για να μπορέσει και το Κοινοβούλιο να αναλάβει το ρόλο που του αναλογεί στη συνέχεια. Με μεγάλη χαρά τους δύο συνεισηγητές θα τους έχουμε πλάι μας και οποιοδήποτε άλλο μέλος της Επιτροπή για να τους εξηγήσουμε καλύτερα τι συμβαίνει και πια πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Οι διαφάνειες που παρουσίασαν οι δύο συνεισηγητές είναι σωστές και ορθές. Υπάρχει μια βασική διαφορά μεταξύ του εργαλείου που υπήρχε αρχικά στο RSP, στο πρόγραμμα στήριξης μεταρρυθμίσεων και το νέο εργαλείο στο BICC. Έχουμε δηλαδή μία ε, συνιστόσα για επενδύσεις και μία συνιστόσα για συγχρηματοδότηση ως εθνικό προαπαιτούμενο. Η κλίδα κατανομής προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τον πληθυσμό, ενώ πρόταση του Συμβουλίου είναι ε, πληθυσμός συν κατακεφαλήν ΑΕΠ. Ε, στόχος είναι περισσότερη συνοχή πάντοτε. Και έχουμε και τη διαδικασία τη διακυβερνητική της διακυβέρνησης για το BICC και αυτό υπάρχει στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δίδεται ε, στρατηγική κατεύθυνση από το Eurogroup στο ε, σύνοδο των κορυφής χωρών μελών της ζώνης του ευρώ Γενικά, παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει επικεφαλής του προγραμμάτους δαπανός και αυτά θέλουμε να τονίσουμε έτσι όπως έχει το κείμενο αυτή τη στιγμή Είμαστε βέβαιοι ότι ο ρόλος μας θα ε, γίνει απολύτως σεβαστός σε σχέση με τις προτεραιότητες για τις δαπάνες. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μπακαρό, νομικό σύμβουλο της ίδιας Γενικής Διευθύνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος εξήγησε τις διαφορές Θέλω να σταθώ σε κάτι, κάτι να προθέσω, προσθέσω. Έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση. Έχουμε την πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο κανονισμό Μιλούμε για το ρόλο του Συμβουλίου της Ζώνης του Ευρώ, το οποίο Συμβούλιο θα καθορίζει τις στρατηγικές κατευθύνσεις, στρατηγικές προτεραιότητες που πρέπει να εξετάζονται από τα κράτη-μέλη και να τα λαμβάνουν υπόψη στην πρόταση του, που υποβάλλουν βάσει του VICC. Δεν είναι όμως ο ρόλος αυτός που έχει να κάνει με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα δαπανών. Εκεί πρέπει να τεθεί ένα όριο μεταξύ του κανονισμού για τη διακυβέρνηση και ε, της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δαπάνες ε, με βάση τα εφιστάμενα κείμενα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκαρικάνο παρακαλώ έχει το λόγο για το Ρινιό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήμουν στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, ε, ε, ε, διαπραγματευόμουν κάτι που μου χρειάστηκε πάνω από 20 λεπτά να το πετύχω. Σας ζητώ συγγνώμη και σας ευχαριστώ για την ευελιξία που δείχνετε να μου δώσετε τώρα το λόγο. Βεβαίως και στηρίζουμε τους συνεισηγητές πρέπει να υπάρξει προϋπολογισμός για τη ζώνη του ευρώ και πρέπει να έχει δυνατότητες και ικανότητες αυτός ο προϋπολογισμός. Η άποψη της Κομισιόν για να λύσει το πρόβλημα της απουσίας κινήτρων και της ιδιοκτησίας των προγραμμάτων ε, από τα κράτη-μέλη είναι κάτι το σωστό και είναι, αποτελεί σωστό σε σημείο εκκίνηση. Γνωρίζουμε πω έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή για τα που κατευθύνεται το Συμβούλιο προ περισσότερη δημοκρατική λόγοδοσία έτσι ώστε να αποσύρονται τελικά ε, θέλουμε εμείς περισσότερη δημοκρατική λογοδοσία. Το Συμβούλιο θέλει να αποσύρονται τα θέματα από το Κοινοβούλιο και να τα εξετάζει το ίδιο μόνο του όλο και περισσότερα και αυτό μας ανησυχεί όλο και περισσότερο. Θα συνεργαστούμε με τους εισηγητές, με όλα τα μέλη και θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια διαδικασία με πιο, που θα είναι πιο δημοκρατική, με μεγαλύτερη λογοδοσία και σε προϋπολογισμό ο οποίος θα είναι αυξημένο και θα ταιριάζει καλύτερα με τις ανάγκες που θεωρούμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ε, τελευταία λόγια και από τους δύο εισηγητές, η Άιντερ Γκαρθία ε, Θαμπάλ. Ευχαριστώ πολύ. Εν συντομία, καταρχάς να ευχαριστήσω τους παριστάμενους Δευτέρα απόγευμα δεν είναι και η καλύτερη μέρα. Ευχαριστώ όλους που ήρθαν και μας άκουσαν. Σημείωσα πολύ προσεκτικά όλα τα σχόλιά σας. Θέλω να διευκρινίσω το εξής. Όταν είπαμε ότι περιμένουμε να έρθει πρόταση της Κροατικής Προεδρίας. Δεν το είπαμε για να ακολουθήσουμε αυτό που προτείνει το Συμβούλιο και το Eurogroup, αυτό είναι προφανές. Λαμβάνοντας υπόψη πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε που παρουσίασε τη θέση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρούμε ότι είναι ε, σωστό να περιμένουμε την πρόταση της Κροατικής Προεδρίας για να μην κάνουμε δουλειά άνευ νοήματος. Άπαξ και μας στείλει το Συμβούλιο την πρότασή του. Με βάση αυτό το έγγραφο εμείς έχουμε το, ως Κοινοβούλιο ε, ελεύθερα τα χέρια, δηλαδή έχουμε κάθε δυνατότητα και ελευθερία να το δεχτούμε, να το απορρίψουμε, να το αλλάξουμε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά δεν έχει νόημα να δουλεύουμε εν κενό, χωρίς δηλαδή να κοιτάζουμε τι κάνουν τα διπλανά, ε, ε τα ε, γειτονικά μας θεσμικά ιδρύματα. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, Υπάρχει ένα θέμα που έχει τεθεί επιτάπητος, δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα παραμείνει, αλλά είναι αρκετά σημαντικό για να το αναπτύξω. Υπάρχει μια ρήτρα ερεσιμότητας σε μακροπρόθεσμη βάση και θέλουμε, θέλουν αυτά τα κονδύλια να τα κλείσουν και να τα συνδέσουν με αυτή τη ρήτρα εκπλήρωσης προαπαιτουμένων σε επίπεδο μακροοικονομίας και σε επίπεδο βάθους χρόνου. Υπάρχει μια φόρμουλα δηλαδή κατανομής. Εμείς ως Κοινοβούλιο όλες οι πολιτικές ομάδες το ξεκαθαρίσαμε, δεν συμφωνούμε με τη χρήση του κριτηρίου του πληθυσμού αποκλειστικά και μόνο για το μηχανισμό της κατανομής. Υπάρχουν διάφορες φόρμουλες που έχουν προταθεί, που βρίσκονται επιτάπητος, όποια και αν υιοθετηθεί τελικά, ε, λαμβάνει περισσότερα υπόψη κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις σε ορισμένα κρατημέλη, ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τα προγράμματα και θα είναι πιο ευπρόσδεκτη από εμάς. Ε, τώρα για τη δίκαιη επιστροφή, για το juste retour που είπαν και οι, προ, οι πράσινοι, ήδη υπάρχει αυτό επιτάπητος. Ανεξάρτητα από το κριτήριο, λέγεται ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει τουλάχιστον να λαμβάνει το 70% αυτού που εισφέρει. Και αυτός είναι ένας τρόπος να διασφαλίσουμε τη δίκαιη επιστροφή και πρέπει να το δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορεί κανείς να διαφωνεί με το σκέλος που έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό ή όχι, όμως θέλουμε να έχουμε ένα πρόγραμμα στήριξης στις μεταρρυθμίσεις για περισσότερες επενδύσεις 7 χρόνια, για 27, χρόνια, ε, για 27 χώρες με 17 ε, ε, δις, δεν νομίζω ότι θα αλλάξουμε και πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να έχουμε ένα εργαλείο σταθεροποιητικό. Ε, ε, κάτι στο οποίο έχουν αναφερθεί και οι δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές επανειλημμένα στο παρελθόν, αλλά μένει πολλή δουλειά να γίνει. Ε, ευχαριστώ. Ο επόμενος συνεισηγητής, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η αρχική μας θέση ως ε, συνεισηγητές ήταν ότι είμαστε ουδέτεροι. Δεν έχουμε ακόμα ετοιμάσει τις απόψεις μα Δεν παρουσιάσαμε αυτά που πιστεύουμε εμείς υπό την ιδιότητά μας ε, πρέπει να αρχάς να εισακούσουμε τους άλλους συναδέλφους και φυσικά να ακούσουμε τι λέει και το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Θα πρέπει λοιπόν να επιδείξουμε ότι τρεις στάση. Προφανώς. Στην παρουσίαση είδαμε τα βασικά κεφάλαια προς συζήτηση και αυτό είναι καλό. Και βλέπουμε και τα σχόλια τα οποία έκαναν οι πράσινοι, το ΕΛΚ, η ΓΚΟΕ, το ΕΣΙΑΡ, και βασικά διαπιστώνουμε ότι η συζήτηση θα πειτρωθεί στα κεφάλαια αυτά. Είναι σαφές. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω στο σημείο αυτό. Σε ό,τι αφορά και αυτά που σχολίασε ο συνάδελφος από την ΚΟΕ, με πολύ διπλωματικό τρόπο αμφισβήτησε το κατά πόσο θα πρέπει καν να υπάρχουν τα εργαλεία αυτά. Ποια είναι η διάκριση μεταξύ των ε, Ταμείων Συνοχής του εργαλείου σύγκλησης και στοπίση. Εδώ τίθεται θέμα έγκυρης ανταπόκριση σε διάφορους εκλεδονισμού Το πρόγραμμα συνοχής ε, προφανώς έχει διαφορετική ε, διαμόρφωση. Σε ό,τι αφορά τώρα το εργαλείο σύγκληση. Ε, μιλάμε για μεταρρυθμίσει, δεν μιλάμε για παρεμβάσει στο επίπεδο τη συνοχή. Μιλάμε για στοιχεία τα οποία πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί, ακόμα και αν τίθεται θέμα βράχει πρόθεσμα. Ολιστική λοιπόν και συνολική μεταρρυθμίση στην ε, παιδεία για το σύστημα εργασία. Αλλά εδώ τέτοια μεγάλα ζητήματα συζητάμε. Φυσικά παραμένουν και τα υπόλοιπα ζητήματα. Είμαστε λοιπόν πολύ ευγνώμονε ε, που ω ε, συνεισηγητέ λαμβάνουμε τα σχόλιά σα. Προφανώ και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με του σκιώδει. Ε, αλλά σε κάθε περίπτωση μην διστάσετε να μα υποβάλλετε σχόλια σε όλη τη διάρκεια τη διαδικασία και να ευχαριστήσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συμμετοχή τη και τη βοήθειά τη. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Το χρονοδιάγραμμα είναι ξεκάθαρο. Η παρουσίαση του σχεδίου εκθέσει θα είναι στις 21 Απριλίου. Και τέλος να αναφέρω την τεράστια καθυστέρηση σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό προοπτική 2021-2027. Θυμάμαι όταν το 2007-2013 ήταν η τελευταία φορά που η συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και μεταξύ των κρατών μελών ήταν ένα χρόνο πιο νωρίς και ακολούθησαν μετά διαπραγματεύσει με το Κοινοβούλιο. Την προηγούμενη φορά η συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων έλαβε χώρα 8 Φεβρουαρίου. Έχουμε μείνει πίσω, είμαστε ακόμα πιο καθυστερημένοι, ακόμα και σε σχέση με αυτό το καθυστερημένο χρονοδιάγραμμα της περασμένη φορές. Αν πετύχουμε τέτοια διακυβερνητική συμφωνία στις 20 Φεβρουαρίου στο Ειδικό Συμβούλιο και φυσικά ποτέ δεν έχουμε πετύχει συμφωνία στην πρώτη, με την πρώτη. Πάντα χρειάζονταν τουλάχιστον δύο φορέ. Α ελπίσουμε λοιπόν να έχουμε θετικό αποτέλεσμα στι 20 Φεβρουαρίου και να ακολουθήσουν οι πραγματεύσει με το Κοινοβούλιο. Ιδάλλως θα είναι τεράστιε οι απώλειε για το 2021 και για το 2022 μάλιστα. Θα πρέπει πάση θυσία να το αποφύγουμε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν τώρα για τι παρεμβάσει σα Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να ξεκινήσει τι κανονικέ τη η Επιτροπή μα.